Συνεχίζετε. Συνεχίζετε συνεδρία συνεδρίε, μοιράστηκαν τα Τα πρακτικά ρωτάω να δω αν υπάρχουν παρατηρήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν παρατηρήσεις, άρα τα πρακτικά θεωρούνται συγκεκριμένα.